του προϊόντος μας για ε, να μπορούμε να τρώμε καλά και να τρώμε υγιεινά. Για αυτό το σκοπό ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ποιότητα και το προϊόντος αλλά της παρέμβασή σας. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο. Πάμε στην επόμενη συζήτηση. Τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά στη συνεδρίαση των G20 εργασίες της Washington 20 και 21 Απριλίου οπότε ας εγκατασταθεί ο πάει τη θέση του κύριου Επίτροπο. Euh, ο κύριος Λάσλο Άντορ λοιπόν έχει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, οι προβλέψεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του ΟΣΑ δείχνουν ότι η ανεργία στις βιομηχανικοποιημένες χώρες εξακολουθούν, εξακολουθεί να αυξάνεται και δεν θα αποκορυφωθεί πριν από το 2011 η ανεργία, το ποσοστό της ανεργίας. Πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες θα κινδυνεύουν να βρεθούν σε ακραία φτώχεια περίπου 1,5 δις θα είναι η φτωχή σε όλο τον κόσμο, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η παρούσα κρίση τόνισε τις επώδυνες αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας. Οπότε υπάρχει συμφωνία ότι χρειάζονται παγκόσμιες δράσεις για να επιληθούν παγκόσμια προβλήματα. Πέρσι στο Pittsburgh οι ηγέτες των G20 υποσχέθηκαν ότι όταν επανέλθει η ανάπτυξη θα, επανέλθει, θα επανέλθει και η απασχόληση. Τούτο λεχθέντος, οι ηγετε g G20 συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για μελλοντική οικονομική ανάπτυξη που αναβάνει υπόψη την απασχόληση. Όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει εδήποτε πλαίσιο δράσεω που θέτουν στο επίκεντρο την απασχόληση, οι ποιοτικέ θέσει απασχόληση, στο επίκεντρο τη ανάκαμψη και βοηθούν τον κόσμο να ξαναβρει δουλειά σε όλο τον κόσμο. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι η απασχόληση είναι, το κατώτατο όριο όσον αφορά, είναι η βάση μάλλον για την ανάκαμψη. Στο Pittsburgh οι ηγέτες κάλεσαν τον Υπουργό Εργασία των ΗΠΑ να συγκαλέσει συνεδρίαση των Υπουργών Εργασία και Απασχόληση των G20. Η εντολή θα είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση της απασχόλησης στον κόσμο και συζητηθούν το πώ οι πολιτικέ απαντήσει στην κρίση επηρεάζουν την όλη κατάσταση και αν χρειάζονται και περαιτέρω μέτρα για την ανάκαμψη. Οι υπουργοί θα πρέπει να δουν μεσοπρόθεσμε πολιτικέ απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμμάτων κοινωνική προστασία και βελτίστων πρακτικών που θα εξασφαλίζει το ότι οι εργαζόμενοι θα ωφελούνται από πρόοδου στην τεχνολογία και στι επιστήμε. Αυτή η συνεδρίαση άνευ προηγουμένου θα λάβει χώρα στη Washington, District of Columbia, στι 20 και 21 Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ισπανική Προεδρία επίση θα συμμετάσχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Διεθνέ Γραφείο Εργασία για την προετοιμασία τη συναντήσεω αυτή, που θα μα προσφέρει, εμά όλου ιδιαίτερω, μια δυνατότητα να προωθήσουμε ε, αξιοπρεπή εργασία σε όλο τον κόσμο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η εφαρμογή των προδιαγραφών του ILO για την επίτευξη του στόχου της βασικής κοινωνικής ασφαλείας είναι κρισίμου σημασίας εδώ να χρησιμοποιηθούν αυτές τις προδιαγραφές. Θα πρέπει η ILO και άλλοι διεθνείς φορείς να αναπτύξουν μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την κατάρτιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στις προσπάθειες μέσω τη νέα πρωτοβουλία για νέε δεξιότητε, για νέε θέσεις απασχόληση. Είναι ένα τμήμα τη πρωτοβουλία για την Ευρώπη του 2020 και ένα πρόγραμμα για νέες δεξιότητες και νέες ε, θέσεις εργασίας. Ποια είναι η βασική πρόκληση, να προχωρήσουμε μια στρατηγική για να αναβαθμίσουμε το εργατικό δυναμικό και να δώσουμε νέε δεξιότητε και να διευκολύνουμε μετά βασία από θέση εργασία σε εργασία και από εκπαίδευση σε εργασία για του νέου. Η εταιρική η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων μπορεί να συμβάλλει τα μάλα Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο κοινωνικό διάλογο και μπορεί να είναι όσον αφορά τη βελτίωση των διαφόρων μέτρων και το σχεδιασμό διαφόρων μέτρων που θα εφαρμοστούν σε διάφορου τομεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμμεριστεί αυτέ τι εμπειρίε με του διεθνεί εταίρου Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί τη επιτευχή σα πρόοδου στη συνεδρίαση στη Washington DC. Οι Υπουργοί Εργασίας των G20 θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε νέα μέτρα τα οποία θα διαμορφώσουν την, το πλαίσιο πολιτικών μετά την κρίση. Αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε ισορροπημένη έξοδο από την κρίση, θέτοντα το επίκεντρο τη ανακάμψεω, την απασχόληση και να ξεπεράσουμε και την κληρονομία τη κρίση. Στόχο είναι να δώσουμε την αναγκαία εισρωή πληροφοριών και προσανατολισμό στου ηγέτε των G20 που θα συνεδριάσουν στον Καναδά και στην Κορέα αργότερα αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει η κυρία Μωρέ Σαρτιέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στα πλαίσια της ε, σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η διάσκεψη αυτή των 20 μας αναγκάζει να διαπιστώσουμε ότι ο πρώτος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των εργαζομένων. Είναι ανάγκη αυτό, γιατί δεν υπάρχει ένταξη στην κοινωνική ζωή αν δεν υπάρχει ένταξη μέσω της επαγγελματικής ζωής. Άρα λοιπόν σήμερα η προετοιμασία στην προετοιμασία της διάσκεψης αυτής ο μόνος στόχος μας πρέπει να είναι καταπολέμηση της ανεργίας. Το είπατε κύριε Επίτροπε ότι η ανεργία έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στον κόσμο ολόκληρο. Όμως βλέπουμε ότι και ανισότητες μεγαλώνουν και μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα μεταξύ των νέων, μεταξύ των ε, εργαζομένων που δεν έχουν μόνιμη δουλειά, μεταξύ των μεταναστών και των γυναικών. Σήμερα 21,4% των νέων είναι στην ανεργία. 14,7% ήταν πριν από δύο χρόνια που ήδη ήταν πολύ Άρα λοιπόν η πρόοδος αυτή καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Πρέπει λοιπόν μαζί να οικοδομήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να βρεθεί υπέρ της ένταξης που να αναγνωρίζει ότι η κοινωνική πολιτική και η πολιτική συνοχής αποτελούν και τον πυλώνα ανάπτυξης της κοινωνίας μας. Θέλω επίσης να επενθυμίσω και το Διεθνές Σύμφωνο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που μας επιτρέπει να βγούμε από την κρίση. Πού βρισκόμαστε όμως σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βασίσει το πλαίσιο της νέας στρατηγικής για μετά το 2010 στην κοινωνική οικονομία των αγορών, την ένταξη και τη διαφάνεια. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εργασίας και Απασχόλησης ελπίζουν να μην ξεχάσουν στη διάσκεψη αυτή ότι μετά θα πρέπει να μιλήσουν για την απασχόληση και για την ε, αύξηση της ανεργίας μπροστά στα εκατομμύρια των ανέργων που έχουν προσθεθεί τελευταία στους ήδη υπάρχοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Επίτροπε, περιμένει από εσά πράξεις για να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τους συμπολίτε μας και να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλεχάνδρο Θέρκας έχει τώρα το λόγο για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι και εγώ πολύ που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα το βράδυ, προετοιμάζοντας την διάσκεψη κορυφής στην Ουάσιγκτον 20-21 Απριλίου. Η κυρία Περβάς Μπερές, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, πολύ θα ήθελε να ήταν εδώ, αλλά λόγω ανώτερας βίας δεν μπορεί να έρθει. Μου έδωσε λοιπόν ε, κάτι που θα σας διαβάσω εγώ στα γαλλικά, στη γλώσσα της και είναι σαν να ακούτε εκείνη. Αγαπητέ Επίτροπε, ενώ η ανεργία στην Ευρώπη ξεπερνάει κατά μεσόρο το 10%, 1,5 εκατομμύρια φτώχοι, η κρίση χτυπάει όλα αυτά τα άτομα. Ήρθε η ώρα λοιπόν κύριε Επίτροπε να δούμε τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και να βάλουμε ως προτεραιότητα την απασχόληση. Χαιρόμαστε για τις εργασίες που έχετε ξεκινήσει και για, τον, για το πνεύμα διαλόγου που έχετε με τους ε, εταίρους σας. Οι ηγέτες κατώ και κυβερνήσεων στο Πίτσβουρκ θέλουν να συνδυάσουν τα μακροοικονομικά στοιχεία με την κοινωνική ανάπτυξη. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ασφάλματα του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην κρίση. Η κρίση όμως ενισχύει τις ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Πρέπει να εμποδίσουμε οι στρατηγικές εξόδου από την κρίση να οδηγήσουν σε καταστροφή του κοινωνικού ιστού. Διότι έχουμε τρία χρόνια τώρα που είμαστε στην κρίση και το βασικό δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, πρέπει να δούμε και την κοινωνική διάσταση της κρίσης. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ο ΩΣΑ, τονίζουν την ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δεν αναφέρεται τίποτα για τον κοινωνικό ιστό στην ιστοσελίδα των 20. Πρέπει όμως να στηρίξουμε την απασχόληση και όχι με τον τρόπο που προτείνεται μέχρι τώρα. Ελπίζω να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Υπουργών Οικονομίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεν θέλουμε τη λογική, τη βραχυπρόθεσμη και θέλουμε η κοινωνική διάσταση να μπει στην καρδιά και των προσπαθειών της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίω. Ευχαριστούμε. Κύριε Σέρκας, το λόγο τώρα η κυρία Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. επιτροπή, συναδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Υπουργή Απασχόληση ε, και Εργασία των ε, G20 καθελούν, όπω ξέρετε, για πολλού ε, εργαζόμενου τα προβλήματα είναι τεράστια. Μειώνεται, μειώνεται το, τα έσοδά δεν υπάρχουν τόσε ε, κατάρτιση Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε να ενισχύονται οι τράπεζες από τα κράτη. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να οδηγήσει σε μείωση των κινήτρων για αποσχόληση. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες και στη χώρα μου, στην Ιλλανδία. Η Κομισιόν λέει ότι ε, είναι καλό που έχουμε τόσο έντονη φορολογική ε, πειθαρχία, αλλά από την άλλη μεριά εμείς χάνουμε πάρα πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει οι θέσεις απασχόληση να είναι το κύριο μέλημα. Τέλος, συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι πολιτικές που είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές του ΑΕΛΟ και θα πρέπει να επιτρέπει η σημερινή οικονομική κρίση να χρησιμοποιηθεί σε μια ε, δικαιολογία για να παρευλεθούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέντο, ένα λεπτό έχει το λόγο ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις ευθύνες που έχουν και εκείνοι έναντι της κοινωνικής κρίσης που είναι σοβαρότατη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνέπεια της χρηματοπιστικής και οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από πλήρη απελευθέρωση των οικονομικών αγορών και στι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου με τρίτες χώρες χωρίς να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται τα συμφέροντα των εργαζομένων και των πληθυσμών. Αυξήθηκε η ανεργία, αυξάνεται η φτώχεια οπότε και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ανεοφιλελεύθερης ε, πολιτικής, της κρίσεω του καπιταλισμού. Στον ΟΣΑ και άλλους διεθνείς φορείς ε, δεν έχουμε πετύχει. Ε, λένε ότι δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο ε, επίπεδο τη ανεργία. Πάνω από 200 εκατομμύρια εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν σε ακραία φτώχεια. Οι φτωχοί εργαζόμενοι μπορεί να φτάσουμε το 1,5 δις. Κυρίως γυναίκες και νέοι θα πληγούν. Ε, θα πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτή τη διαδικασία ε, της μείωσης των κοινωνικών προδιαγραφών εργασίας θα πρέπει να είναι ποιοτικέ οι θέσει απασχόληση, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, αν μη τι άλλο να σεβόμαστε τι προδιαγραφέ του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Αν δεν σεβαστούμε αυτές τις, ε, αυτά τα κριτήρια, θα μπορούμε να βγούμε την κρίση. Ευχαριστώ, κυρία Φιγκεραίδο. Και τώρα επόμενο γυμνητή, κύριο Γκόντ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Γκόντ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, για μας όλους είναι πολύ ευχαριστώ ότι στο γύρο των G20 συναντώνται οι Υπουργοί Εργασίας και έτσι μπορούν να θεωρηθούν ισότιμοι των Υπουργών Οικονομικών. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ποτέ ένα παράδειγμα στο οποίο ε, σε μια διεθνή οικονομική κρίση υπάρχει μια τέτοια υπουργική συνάντηση για να εξεταθούν τα προβλήματα των εργαζομένων. Σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί φαίνεται ότι η οικονομική πίεση της κρίσης μειώνεται, από την άλλη μεριά αυξάνεται η ανεργία και η ένδια και γνωρίζουμε ότι αυτό θα έχει μακροπρόθεσμα κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε να εξαπλώνεται ο εξτρεμισμός και αυτό σημαίνει ε, μια, έναν κίνδυνο μακροπρόθεσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι πολιτικοί να προετοιμάσουν κάποιους ε, κανόνες για να μπορέσει να μειωθεί η ένδια, να αυξηθεί η απασχόληση. Ε, α, η μικροχρηματοδότηση είναι θέμα που θα ζητηθεί ε, G20. Είναι από την άλλη μεριά λυπηρό ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να χρωμοδοτήσει για τη συνάντηση αυτή και μπορούμε μόνο προφορικά να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λίν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έπληξε τους απλούς ανθρώπους πάρα πολύ σκληρά η οικονομική κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε θετικά αποτελέσματα από τη συνεδρίαση προεργασίας των G20 το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ζητήθηκε, αναφέρθηκε. Και ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Χαίρομαι ότι θα επικεντρωθούν μόνο στο χρηματοδοτικό τομέα. Θα εξετάσουν τι κοινωνικέ συνέπειε τη κρίση. Έχει σπάσει ρεκόρ η ανεργία σε πολλέ χώρε στον κόσμο. Πρέπει να δούμε πώ μπορεί να επιστρέψει ο κόσμο στι δουλειέ του. Πραγματικέ θέσει ασχαδίε. Προγράμματα κατάρτιση θα πρέπει να είναι καλά. Να καλύπτουν τι ανάγκε τη στιγμή να βρούμε βέλτιστες πρακτικές από χώρες που ήδη έχουν θεσπίσει μέτρα. Πρέπει να εξεταστούν και να μεταφερθούν οι καλές πρακτικές σε άλλες χώρες. Να βοηθήσουμε τους πιο περιθωριοποιημένους ανθρώπους της κοινωνίας. Έγινε δουλειά σε άλλες χώρες. Γιατί να μην μάθουμε. Θα πρέπει βασικέ βασικές συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές. Και η Σύμβαση ΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων ανθρώπων να γίνονται σεβαστά. Εκείνοι που δεν προστατεύονται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προστατευτούν στο μέλλον. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Λίν. Ο κύριος Τόμας Χάντελ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η διάσκεψη του G20 στο Πίτσκου έδωσε καλά, ε, καλές οθήσεις γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόληση και να δέδωσε προτεραιότητα στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ε, πιέσουμε τα μέλη του G20 να μην μειώσουν τις ε, ενισχύσει που δίνονται. Δεύτερον, να εισαχθεί περιορισμένη χρόνου εργασία για να μην απολυθούν οι θέσεις απασχόλησης και δεύτερον να προωθήσουν την αηφόρο οικολογική ανάπτυξη και τέλος να ε, προωθήσουν μέτρα διασφάλισης πράγμα που εξασφαλίζει και την αγοραστική αξία στην εσωτερική αγορά και καταπολεμά την ένδια. Η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι Υπουργοί Εργασία στην Ευρώπη για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον κοινωνικό διάλογο, όπω θέλει και ο Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χέντελ. Η κυρία Σιλβάνα Ράπτη. Ένα λεπτό. Parfait. Merci. Merci bien. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ουάσιγκτον στις 20 Απριλίου θα έχουμε μία πρεμιέρα. Για πρώτη φορά θα συνεδριάσουν Υπουργοί Απασχόλησης των 20 περισσότερο πλούσιων περιοχών της γης. Εκεί η φωνή της Ευρώπης πρέπει να ακουστεί πάρα πολύ δυνατή. 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν στην ευρωπαϊκή περιοχή την τριετία που έρχεται και αυτό θα έχει επίπτωση στην ανάπτυξη θα τραυματίσει την κοινωνική συνοχή θα προκαλέσει κοινωνικές αναταράξεις. για την ευρώπη η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. είναι επιτακτική ανάγκη να τεθούν στόχοι. Ρεαλιστική, συγκεκριμένη, μετρήσιμη, στόχοι μακροπρόθεσμοι και άμεση. είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους πολίτες της ευρώπης αξιοπρεπή εργασία. είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούμε να διασφαλίζουμε τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. κοντεύουμε να ξεχάσουμε το αυτονόητο ότι η εργασία είναι μοχλός ανάπτυξης. επιτέλους νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομική πολιτική χωρίς να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας την παράμετρο απασχόληση. κλείνω κυρία πρόεδρε λέγοντας ότι διαφορετικά αντί να μιλάμε για συμβούλιο υπουργών απασχόλησης θα μιλάμε για συμβούλιο υπουργών ανεργίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση για την ανεργία αν δεν αλλάξει και δεν αντιστραφεί η σημερινή λογική όπου δίνουμε προτεραιότητα στο κεφάλαιο και όχι στην εργασία. Χωρίς νέα κατανομή του πλούτου που σημαίνει αύξηση των μισθών και της κοινωνικής προστασίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ανάκαμψη, κοινωνική πρόοδο που είναι αναγκαία για την έξοδο από την κρίση. Οι 20 πρέπει να φροντίσουν να κινητοποιήσουν ε, το διεθνή τραπεζικό τομέα για να εξυπηρετήσει την απασχόληση, τους μηχανισμούς που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και να δημιουργηθεί μια νέα οικονομία υπέρ του περιβάλλοντος. Συγχρόνως, η κίνηση των κερδοσκοπικών κεφαλίων πρέπει να αλλάξει και να ενισχυθεί η εργασία. Χρειάζεται κατάρτιση για να προετοιμαστούμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και έτσι θα οδηγηθούμε σε μια νέα βιώσιμη οικονομία. Ευχαριστούμε. Συνάδελφε Λιαρίκ, τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch Η συνάδελφος Τικά έχει πρώτο το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί υπότροπε ηγέτες των G20 το Δεκέμβριο του 2009 αποφάσισαν κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή να διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης και να δημιουργηθούν νέες. Στις προγνώσεις όμως του Διεθνού Γραφείου Εργασίας για την Ανάπτυξη 3%, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ και του Διεθνούς, και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δείχνουν ότι θα αυξάνεται η ανεργία μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2011. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχαν αρνητικές συνέπειες επί των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επί των προπολογισμών των κρατών μελών. Οι Υπουργοί Απασχόλησης των G20 θα πρέπει να ζητήσουν να δοθεί υποστήριξη στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολία και αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να χορηγείται μέχρι ότου να έχουμε μείωση της ανεργίας. Θα πρέπει να βρουν οι Υπουργοί μέτρα για να υποστηρίξουν τους δημοσίους υπαλλήλους και εκείνους που πληρώνονται από δημόσιους πόρους, από γιατρούς, δασκάλους που χάνουν τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Η έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, διότι για πρώτη φορά οι Υπουργοί Εργασία των G20 συνεδριάζουν και απασχόληση. Μετά από τη συνεδρίαση στο Pittsburgh των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των G20, εκεί είχαν συμφωνήσει ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα το θέμα τη διατηρήσεω των θέσεων απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Δυστυχώ επιδεινώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση και, και σε κάποια κράτη-μέλη έφτασε σε κρίσιμα επίπεδα το ποσοστό της ανεργίας και και επιδεινώνεται η κατάσταση διότι τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν είναι σωστά. Και γιατί κυρίως πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στους G20 θα πρέπει να τονιστούν ειδικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Υπάρχει φόβος στους ανθρώπους, υπάρχει απαγοήτευση και αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, η Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Πράγματι, νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι Υπουργοί Εργασίας και Απασχόλησης των G20 συνεδριάζουν και προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις. Πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία, πώς θα δημιουργηθούν έτσι θέσεις εργασίας. Η κατάσταση είναι περιπλοκότατη Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,5 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι. Και αυξάνεται ο αριθμό των ανεργών παντού. Στη πατρίδα μου, στη Λιθουανία, 300.000 άνθρωποι είναι οι επίσημα καταχωρημένοι άνεργοι. Τα 20 χρόνια τη ανεξαρτησία αυτό είναι πρωτάκουστο. Είναι σημαντικό λοιπόν όπου οι Υπουργοί Εργασία των G20 θα ελέγξουν τη θέσπιση ειδικών μέτρων όχι μόνο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, καλά αμοιβωμένων θέσεων εργασίας, που οδηγούν σε αξιοπρεπή επιβίωση, διαβίωση μάλλον, και όχι φτώχεια. Χαίρομαι που τελικά θα κατέξω σε κάποιες αποφάσεις. Ευχαριστώ λοιπόν τη διαδικασία εδώ του Κασάη και θέλω να δώσω τον, το λόγο στον Επίτροπο Αντόρ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έγινε η συζήτηση αυτή σήμερα πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Εργασίας ε, και Κοινωνικών Υποθέσεων στην του G20 και δεν είναι η, πρώτη, η μόνη διάσκεψη για την οποία θα ακούσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και μια άλλη διάσκεψη κορυφής ε, που είναι πιο νωρίς και θα πρέπει να ακούσει τι έχετε να πείτε σήμερα. Έχω κατά νου ποιες αύριο εδώ στις Βρυξέλλες που θα είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει την ημερησία διάταξη, την ατζέντα του 2020 για να προωθήσει την απασχόληση και να μειώσει την ένδια. Σημαντικοί στόχοι που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει νομίζω να ε, εκτιμήσουμε ότι η διεθνή οικονομία βρίσκεται σε κρίση εδώ και δύο χρόνια και αυτό δεν είναι θέμα μόνο στατιστικών. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Γκέντς ε, ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε και τον πολιτικό κίνδυνο, το κίνδυνο δηλαδή που παρουσιάζει αυτή η κρίση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ελπίζω ότι οι ηγέτες που θα συναντηθούν αύριο θα κατανοήσουν αυτό το θέμα και θα καταλήξουν σε υπεύθυνες, ε, συμπεράσματα. Ενώ είναι δύσκολο να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες σε όλο τον κόσμο και ήταν δύσκολο να προωθήσουμε αξιόπιστα τη δέσμευσή μας για την αντιμετωπίση τη ε, ένδυας και τη ανεργία μέσα στα φρέσια του G20. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον έχουν απογαλακτιστεί από τους υπουργού οικονομικών, έχουν χειραφητηθεί από αυτούς και κατά πόσον θα μπορέσουν πραγματικά να αποφασίσουν κάτι και όχι να ανταλλάσσουν απλώς απόψεις. η δημοσιονομική ισχύ των κρατών έχει εστιαστεί στην υποστήριξη των τραπεζών. Αυτό ήταν η κύρια προτεραιότητα μέχρι στιγμής, αλλά τώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στην δημιουργία απα... θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική που δεν υποσκάπτει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή το δυναμικό επένδυσης θα πρέπει να υπάρχει η τάξη, να αυξηθεί η σταθερότητα και να μην υπάρχει τόση πίωση στα κρατη να κάνουν περικοπές παράλογες που θα έχουν επιπτώσεις στην απασχόληση. Συμφωνώ ότι ο ακρογωνιαίος ε, λήθος για τα πρότυπα αυτά είναι το Διεθνές ε, Γραφείο Εργασίας, το ΑΕΛΟ. Υπάρχουν και πάρα πολλά πρότυπα που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές σχέσεις. Το πλαίσιο των, της ομάδας των 20, του G20, είναι σημαντικό για τις συζητήσεις ανά τον κόσμο, όχι μόνο για τις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά και για θέματα δημοσιονομικά και για θέματα όσον αφορά παραδείγματο χάρη το φόρο στις ε, ε, συναλλαγές που συζητιέται που και που. Ε, είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους που μίλησαν και θα μεταβιβάσω το μήνυμά σας στους άλλους εταίρους στην ε, G20. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ σας ευχαριστώ Επίτροπη κυρία Άντορ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος. Το επόμενο σημείο της διάταξης είναι η δήλωση της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Μπορούμε να χαιρετήσουμε.